Συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Μετά από την συναρπαστική αυτή συνεδρίαση με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, σας ζητώ να θρέψουμε την προσοχή μας σε πιο τεχνικά ζητήματα της Επιτροπής ΣΕΝΤΕ. Είναι τεράστια η αίθουσα για την υποεπιτροπή μας, αλλά τι να κάνουμε, θα τα βγάλουμε πέρα. Επιτρέψτε μου να ακολουθήσουμε την ημερήσια διάταξη της σημερινής συνεδρίασης, μετά από κάποιες αλλαγές που έγιναν, σε ό,τι αφορά την ε, σειρά. Να εγκρίνουμε τα πρακτικά των τελευταίων συνεδριάσεων, της τελευταίας συνεδρίασης. 22 Μαρτίου και 23 Μαρτίου. Μέχρι το τέλος της σημερινής συνεδρίασης έχετε χρόνο. Σε περίπτωση που έχετε σχόλια, επιφυλάξεις για τα πρακτικά. Αν δεν υπάρχουν σχόλια θα θεωρηθούν εγκεκριμένα. Το επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης είναι η δεύτερη εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης για τη στρατηγική της Ευρώπης για το διάστημα. Η συγητής, ο κ. Τζέφρι Φανόρντον. Δυστυχώς. Κολλείται και δεν μπόρεσε να παραβρεθεί σήμερα. λόγω σημαντικών ανελημμένων υποχρεώσεων στην περιφερειά του. Ζητά συγγνώμη από όλους τους παρόντες. Στείλαμε ένα σημείωμα προς όλα τα μέλη. Το έστειλε γραμματεία, αν δεν κάνω λάθος. Παρακαλώ λοιπόν να ελέγξετε τα email σας για να διαβάσετε τα σχόλια του κυρίου Φανόρντεν. Ζητώ συγγνώμη εκ μέρους του. Και τώρα θα ήθελα να καλέσω τους παρόντες και ότες συζητητές, αν συμφωνούν, να επεξεργαστούμε παρόλα αυτά το θέμα αυτό. ο κύριος Βανόρντον θα διοργανώσει συνάντηση των σχεδόν για την εξέταση των τροπολογιών. Ζητώ λοιπόν από τους σκιώτες να κάνουν σχόλια. Το ΕΛΚ εκπροσωπείται από τον κύριο Στροβιεύσκη. Αν θέλετε να πάρετε το λόγο, παρακαλώ αγαπητέ συνάδελφε, για να μας παρουσιάσετε τα σχόλια επί της νομοδότησης projektu pana e, Tak, oczywiście, pani przewodnicząca. Ναι, βεβαίω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο και είναι πολύ ατυχέ που δεν είναι παρόν σήμερα εδώ ο κύριο Φανόρντον. Αυτό που είναι εξαιρετικό φυσικά είναι η έκθεσή του, η γνωμοτότησή του. Πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο το περιμέναμε εδώ και καιρό και το οποίο υποστηρίζουμε σε μεγάλο βαθμό. Δεν κατατέθηκαν και πολλές τροπολογίες, 36 μόνο. Οι πιο πολλές εξ αυτών δε είναι αποδεκτές από την ομάδα μου. Ω εκ τούτου θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι με ένα έγγραφο το οποίο καταρχάς είναι πάρα πολύ απαραίτητο. Η δουλειά του κ. Φανόρντεν εδώ δεν είναι μόνο αποδεκτή αλλά και πραγματικά πολύ ποιοτική. Τον ευχαριστούμε. Κάποιες παρατηρήσεις τώρα και κάποιες λεπτομέρειες να σχολιάσουμε. Αυτή η γνωμοδότηση αποτελεί μια εξαιρετική βάση για τις περαιτέρω συζητήσει. οι οποίε θα είναι στρατηγικής σημασίας. και θα αφορούν και πάρα πολλά συγκεκριμένα στοιχεία. Είναι πάρα πολύ λοιπόν σημαντική η γνωμοδότηση αυτή σε ό,τι αφορά τα τεχνικά συγκεκριμένα επιμέρου στοιχεία. Πέραν τούτου, υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις οι οποίες συναντιόνται αφενός παραμελούνται διάφορες διαστημικά επιχειρήματα, εγχειρήματα τα οποία ε, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για σκοπούς ασφάλειας, αλλά από την άλλη υπάρχει και μία αντίστροφη τάση. Τα κράτη-μέλη να κάνουν τα δικά τους ε, και να μην υπάρχει συντονισμό με το ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά το κόστο, τι δαπάνε, σε ό,τι αφορά και το δυναμικό ανάπτυξη. Θεωρώ λοιπόν ότι πολλά μπορούμε να κάνουμε από κοινού στο σημείο αυτό για να βελτιώσουμε στο σύνολό τη την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Τα συστήματα αυτά δεν μπορούν όμω να είναι υψηλή ποιότητα στα συστήματα, δηλαδή σε ό,τι αφορά την διαστημική τεχνολογία. Δεν μπορούν να είναι υψηλή ε, ποιότητα αν δεν υπάρξει συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα χρειαζόμαστε μια κοινοτική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τα δορυφορικά συστήματα, προκειμένου να είναι η καλύτερη δυνατή η ποιότητα των συστημάτων αυτών που θα αναπτύξουμε και έτσι να ενισχύσουμε και την ασφάλεια των συναδέλφων, των πολιτών μας. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, και να αναφέρει στο σημείο αυτό ότι η αρμόδια επιτροπή είναι προφανώς η Επιτροπή Βιομηχανίας. Η Επιτροπή Ήτρε και δικός μας ρόλος είναι η γνωμοδότηση, η χορήγηση γνωμοδότησης. Η Φροντζούλη, από και <clears throat> Ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ασφαλώ είναι πολύ σημαντικό. Θα ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε μαζί μα την Κρυφανόρδεν, Όρδεν. Αλλά καταλαβαίνουμε την κατάσταση. Προτείνουμε λοιπόν και εμεί να αποστείλουμε με email τα σχόλιά μα προ την Κρυφανόρδεν, Αλλά ασφαλώ, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να υποδείξω και εγώ κάποια ζητήματα τα οποία α, έχουν να κάνουν με το πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Λαμβάνοντα υπόψη ε, την, ε, το ευάλωτο των δυστημικών αυτών συστημάτων από κρατικούς, σε επιθέσεις από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς, θα ήθελα να, να υπογραμμίσω επ' ότι το διάστημα είναι κρίσιμη σημασία για την ασφάλεια μας και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει αυτονομία και ασφάλεια σε ό,τι αφορά αυτές τις υπηρεσίες μας που βασίζονται στο διάστημα. Επίσης, τονίζεται στην γνωμοδότηση ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες με μεγάλη εξουσία που μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο. Άρα θα πρέπει να εξετάσουμε πώς μπορούμε να βρούμε κοινούς κανόνες για να είναι το διάστημα ασφαλές και προσβάσιμο σε όλους. Ε, συμφωνώ ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας στο διεθνές προσκήνιο και υπάρχει συνεργασία από την άποψη αυτή με τις, τα κράτη του ΝΑΤΟ, με την Ιαπωνία, για να υπάρχουν κοινά να προσπιστούν τα κοινά συμφέροντα. Θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει ο κλάδος από ευρωπαϊκή άποψη να μπορεί να τροποποιείται σε μια ταχεία μεταβαλλόμενη κατάσταση σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην ασφάλεια, για παράδειγμα. Επίση, πιστεύω ότι οι διμερεί σχέσει μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και των ΗΠΑ στα θέματα αυτά θα πρέπει να καλύπτει και τι καταστάσει ε, που αφορούν την ασφάλεια ανταπόκριση σε διάφορες καταστροφές, ε, έλεγχος όπλων, τρομοκρατικές επιθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσία Διαστήματος θα πρέπει να δράσει από κοινού με τη βιομηχανία για να προασπίσει τα, δικαιώ, τα συμφέροντά της στο διάστημα. Να τονίσουμε επίσης ε, ότι είναι σημαντική η ανάπτυξη της τεχνολογίας ε, διαστήματος καθώς και η ανάπτυξη συστηματών διπλής ε, χρήσης ε, όπως γίνεται σε διάφορα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να προωθηθεί αυτή η διπλή χρήση και να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ της υπηρεσίας τοπικής δράσης, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνα, του Ευρωπαϊκού Τροφορικού Κέντρου και των κρατών μελών. Σας ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος και ο που να θέλει τον λόγο. Ο κύριος που είναι ε, η κυρία Λόζινγκ που είναι υπεύθυνη από πλευράς Γκουε μόλις εγκατέλειψε την αίθουσα. Νομίζω ότι έτσι μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Προφανώς η συνάντηση μεταξύ των σκιωδών συγητών θα είναι απαραίτητη και ο κ. Φανόρντεν θα τη συγκαλέσει σύντομα προκειμένου όλα να γίνουν σύμφωνα με τους τύπους. Η ψηφοφορία στην ΑΦΕΤ θα γίνει στις 30 Μαΐου και στην Ολομέλεια θα ψηφιστεί η έκθεση. Α, πρώτα θα, το θέμα θα περάσει στην Ήτρε στις 22 Ιουνίου και δεν ξέρουμε σε ποια ολομέλεια τελικά θα ψηφιστεί. Θέλω τώρα να κάνουμε μια μικρή διακοπή ο υπονάβαρχος ε, ε, είναι κάπου εδώ κοντά το γνωρίζουμε αυτό ο... Ε, σε λίγο θα είναι μαζί μας μαζί με τον κύριο Γκος κάνουμε μια μικρή διακοπή να προετοιμάσουμε τα έδρανα και θα περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Uh, Παρακαλώ, λάβετε θέση. Ξεκινάμε το τελευταίο σημείο, σημείο της σημερινής ημερησίας Αύριο σας θυμίζω ότι ε, θα συναντηθούμε το πρωί ξανά με αλλαγή στην αίθουσα σημειώστε την καινούργια αίθουσα, έτσι μην την κάνετε λάθος. Περνάμε στις, ε, το πρόγραμμα ανάπτυξης ε, δυνατοτήτων και την ε, εξέτασή του. Καλωσορίζω τον κύριο Ρίνι Γκος, υποδιευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας και τον υπονάβαρχο Βάλτεμαρ Γκλούσκο, ε, υποδιευθυντή, ε, μάλλον υπαρχηγό του Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Επιτελείου Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Θα δώσω καταρχήν το λόγο στον κύριο Γκος. Ε, Ευχαριστώ κύριε Αφωτίγα Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ για να σας ε, παρουσιάσω ένα από τα ε, πιο σημαντικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το CDP, όπως το ονομάζουμε, το Πλάνο Ανάπτυξης Δυνατοτήτων. Καταρχήν, γιατί το CDP είναι τόσο σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα επίπεδα. Μετά θα σας εξηγήσω λίγο το ιστορικό και τις ε, βασικές λειτουργίες του CDP ε, τι καινούργια στοιχεία θέλουμε να προσθέσουμε στην αναθεώρησή του και ε, θα σας μιλήσω για τις ε, προτεραιότητες που θα προκύψουν στο τέλος της αναθεώρησης το 2018. Όπως γνωρίζουμε, το περιβάλλον ασφάλισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αλλάξει τα τελευταία δύο χρόνια. Στην Ευρωπαϊκή Παγκόσμια Στρατηγική αναφέρεται ότι περνάμε περίοδο υπαρξιακή κρίσης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι οι και φορείς, συμπεριλαμβανομένης και τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτέ τι κοινέ προκλήσει. Και το e CDP θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο ευρύ πλαίσιο των προτεραιοτήτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πρωτοβουλίων τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για μια πιο αποτελεσματική άμυνα. Ε, η συνολική σφαιρική στρατηγική λέει ότι το, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει το CDP και, τις, ε, ε, και να αποτελέσει το πρόγραμμα αυτό μια σύνδεση ανάμεσα στην δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή της Κομισιόν. Τα κράτη-μέλη έχουν συμφωνήσει ε, να καταστήσουν πιο σαφείς τις προτεραιότητες σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές δυνατότητες μέσω της αναθεώρησης του CDP. Τέλος, το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Άμυνας αναφέρεται στο CDP λέγοντας ότι οι πρωτοβουλίες του προγράμματος αυτού ε, θα, οι πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ωφεληθούν από το CDP. Συνεπώς το CDP θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών στρατιωτικών ικανοτήτων. Τι αφορά όμως. Το CDP είναι ένα σχέδιο που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να θέσουν προτεραιότητες για την εργασία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας. Ε, στηρίζει την ανάπτυξη των αμυντικών ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της στρατιωτικής συνεργασίας. Δεύτερον, ε, προωθεί την τεχνολογία και την στρατιωτική έρευνα, ενισχύει την στρατιωτική ε, ε, βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωσης και αποτελεί ενδιάμεσο με τις, ευρωπαϊκές, με τις άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές. Βασικός στόχος του CDP είναι να δημιουργήσει ένα πανόραμα στρατιωτικών απαιτήσεων μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. βασίζεται σε μια σειρά από input όπως τα, τα σχέδια ανάπτυξη των κρατών μελών, την ανάλυση των τεχνολογικών δυνατοτήτων και προκλήσεων για το μέλλον, καθώς επίσης και ε, την άποψη της στρατιωτικής βιομηχανίας. Ε, όλες αυτές οι πληροφορίες ε, πρέπει να τύχουν επεξεργασία έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια συνολική εικόνα. Επί τη βάση αυτής της εικόνας είναι δυνατόν να εντοπιστούν συγκεκριμένες προτεραιότητες και δράσεις που χρειάζονται. Ταυτόχρονα το σχέδιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σημείο αναφοράς για ε, τους διάφορους ενδιαφέρουσες φορείς και αυτούς που λαμβάνουν ε, αποφάσεις ε, σε εθνικό επίπεδο. Οπότε το CDP οδηγεί σε μια πλήρη εικόνα των στρατιωτικών δυνατοτήτων και θα αποτελέσει εργαλείο σε εθνικό επίπεδο και για τις επιχειρήσεις που θα βρουν καινούριες ευκαιρίες, αλλά και για αυτούς που θα θέσουν προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο για το σε ποιο τομέα θα πρέπει να αναπτυχθούν οι ε, στρατιωτικές ικανότητες. Με αυτόν τον τρόπο το CDP αποτελεί εργαλείο ενημέρωσης, ε, εντοπίζει τομεί στου οποίου μπορεί να βελτιωθεί η συνεργασία μέσο πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και καθώς επίσης εντοπίζει και συγκεκριμένες κοινέ προτεραιότητες ε, σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές ε, δραστηριότητες εφαρμογής του. Οπότε το CDP ενισχύει, διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και στηρίζει την διαδικασία ανάπτυξης ε, ικανοτήτων από τον προγραμματισμό μέχρι την εφαρμογή και την υλοποίησή τους. Τώρα, τι το καινούριο έχει αυτή η αναθεώρηση. Το πρώτο CDP υιοθετήθηκε το 2008, ενημερώθηκε το 2011 και τροποποιήθηκε το 2014. Ε, από τον Νοέμβριο του 2016 οι Υπουργοί Άμυνα ε, ζήτησαν όχι μόνο να ενημερωθεί το CDP αλλά να αναθεωρηθεί με καινούριες προτεραιότητες μέχρι την άνοιξη του 2018, λαμβάνοντα υπόψη το καινούριο στρατηγικό πλαίσιο. Κατόπιν αυτών των κατευθύνων αμών, ήδη από το 2016 ξεκινήσαμε να αναθεωρούμε το περιεχόμενο του CDP με μια καινούρια μεθοδολογία εν μέρη. Η επόμενη εκδοχή του για πρώτη φορά ε, θα, ενταχ, θα συνενωθεί με τα συμπεράσματα από ασκήσεις που έχουν γίνει, για παράδειγμα εναντίον των κινδύνων του κυβερνοχώρου ε, που έχουμε κάνει ε, και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπόλ, ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης, το ΝΑΤΟ κλπ. Οι ασκήσεις αυτές θα επηρεάσουν κατά πολύ τις καινούριες προτεραιότητες του CDP. Το CDP επίσης κοιτάει και μακριά, μακροπρόθεσμα. Υπ' αυτή την έννοια θα κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου έτσι ώστε να, να εντοπίσουμε ε, τις ε, μελλοντικές ε, τάσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τα εθνικά προγράμματα. τι πρέπει να κάνουμε τώρα για να είμαστε έτοιμοι για το μέλλον. Επιπλέον, το επόμενο CDP θα λάβει υπόψη τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Στρατιωτικής Επιτροπής που θα είναι πολύ ρεαλιστικές σε ό,τι αφορά την εκτίμησή τους. Τέλος, εκτός από τις εθνικές απόψεις, για πρώτη φορά θα λάβουμε υπόψη και την ε, κοινότητα έρευνας και τεχνολογίας ε, ε, που θα μας επιτρέψει να παρακολουθήσουμε τις τεχνολογικές εξέλιξεις και έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη και τις ανάγκες και απαιτήσει που η τεχνολογική εξέλιξη δημιουργούν σε μας. Τώρα, πρωτοβουλίε, ε, προτεραιότητε, συγγνώμη, που προκύπτουν από τη CDP. Οι προτεραιότητε θα τύχουν συμφωνίε μεταξύ των κρατών μελών του χρόνου. Και θα διαφέρουν από τι σημερινέ προτεραιότητε ω εξή. Θα διαφέρει το πεδίο του, που θα έχει σχέση με τι πιο επίκαιρε δραστηριότητε τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτή την έννοια το CDP θα αποτελεί σύνδεσμο ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα αλλάξει ε, ο εστιασμός, η εστίαση, ε, θα εστιάσουμε πιο πολύ στη συνεργασία, ε, θα εξετάσουμε ε, τις αδυναμίες αυτή τη στιγμή, τις απαιτήσει μεσοπρόθεσμα και τις ευκαιρίες στο μέλλον. Θα πρέπει να δούμε όλες τις σχετικές διαστάσεις, έρευνα ανάπτυξη, κοινή, κοινές αγορές, απαιτήσεις, κοινές απαιτήσεις και προδιαγραφές για συγκεκριμένα σχέδια κλπ το, αυτά, αυτές οι απαιτήσει θα καθοριστούν από κοινού μεταξύ των κρατών μελών, της, ε, του κλάδου κλπ. Τέλος, οι προτεραιότητες θα είναι πιο σημαντικές και για τη βιομηχανική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να συνδέσουμε αυτές τις προτεραιότητες με τους ε, ενδιαφερόμενους ε, εμπλεκόμενους φορείς όσο πιο νωρίς γίνεται. Είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια στρατηγική αυτονομία. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να έχουμε και μια ισχυρή τεχνολογική και βιομηχανική βάση. Χωρίς αυτήν τα κράτη-μέλη θα εξαρτώνται από τρίτους. Πρέπει να, υπογράψω, να υπογραμμίσω ότι η περιπλοκότητα της αλυσίδας ε, παραγωγής ε, δεν μας επιτρέπει να είμαστε 100% αυτόνομοι και να βασιστούμε μόνο στα κράτη-μέλη. Όμως είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ελευθερία δράσης και αποτελεσματικότητα. Αυτό σημαίνει και ανάπτυξη δικών μας εξαιρετικών ικανοτήτων. Συνεπώς οι προτεραιότητε του CDP θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις τεχνολογίες, τις ικανότητες παραγωγής και ε, τις ε, ε, ε, ε και, και τεχνολογικές ικανότητες που διαθέτουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, να υπογραμμίσω ότι ο στόχος του CDP και των προτεραιοτήτων του είναι να στηρίξουμε καταρχήν τα κράτη-μέλη στις προσπάθειές τους να αναπτύξουν συνεργατικές ικανότητες. Δηλαδή, οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσία Άμυνα είναι αποτέλεσμα συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών. Αυτές όμως οι ικανότητες θα είναι ικανότητες των κρατών μελών, θα είναι πόροι και περιουσιακά στοιχεία των κρατών μελών που θα αποφασίζουν κατά το δοκού να τα χρησιμοποιούν ή όχι. Επειδή είναι μάλιστα και οι περισσότερε χώρε είναι και σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, ε, θα... οι ικανότητε αυτέ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε επιχειρήσει του ΝΑΤΟ. Συνεπώ, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ωφελείται άμεσα, το ΝΑΤΟ θα ωφεληθεί επίση έμεσα. Εφόσον τα κράτη-μέλη θα αναπτύξουν τι ικανότητέ του και θα μπορέσουν να συνεισφέρουν στην κοινή ασφάλεια όλων. Αντιστρόφως και το CDP επωφελείται από την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Τα κράτη-μέλη όμως θα το εφαρμόσουν. Για παράδειγμα, τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ε, Άμυνας είναι, μπορούν να αποφασίσουν να καλέσουν την ε, Υπηρεσία Άμυνας σε κοινέ συνεδριάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ έτσι ώστε να την εμπλέξουν και να είναι δυνατόν να η υπηρεσία ε, ε Ευρωπαϊκής Άμυνας ε, να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα. Αλλά και αντιστρόφως, το ΝΑΤΟ μπορεί να συμμετάσχει ως παρατηρητής σε ασκήσεις εναντίον απειλών του κυβερνοχώρου που λαμβάνουν χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτόν τον τρόπο τα κράτη-μέλη μπορούν να εξασφαλίσουν μια λογική συνέχεια ανάμεσα στις δράσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς άλλες Ε, Αυτό είναι ένας από τους στόχους αναθεώρησης του CDP. Όμως, να υπογραμμίσουμε ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι η κατευθυντήρια αρχή. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον καθεσμό των προτεραιοτήτων. Τελειώνοντας να πω το εξή. Το αναθεωρημένο CDP του 2018 θα λαμβάνει υπόψη τους στόχους των νέων στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών. Ε, και παρόλο ότι ε, ε, είναι εστιάζει στις ικανότητες, στις στρατιωτικές ικανότητες, θα δημιουργήσει μια καλύτερη εικόνα των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο και δεν θα απευθυνθεί μόνο στους ε, υπεύθυνους λήψη των αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο, αλλά και στη βιομηχανία και στα ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα. Οι προτεραιότητες ανάπτυξης στρατιωτικών ικανοτήτων θα στηρίξουν καλύτερα τη δράση των κρατών μελών και θα διευκολύνουν την ένταξη της ευρωπαϊκής διάστασης στις, ευρωπαϊκές, στις εθνικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Ε, δηλαδή θα είμαστε πιο πολύ εστιασμένοι σε εθνικό επίπεδο στις ε, κοινωνικούς ευρωπαϊκούς στόχους. Ευχαριστώ. Τώρα ο υπονάβαρχος Γκλούσκο, υποδιευθυντής του Στρατιωτικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Στόχος της παρουσίασής μου είναι να σας καταδείξω τον ρόλο που παίζει το επιτελείο του στρατού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα επικεντρωθώ στην Στρατιωτική Επιτροπή. Θα αναπτύξω λίγο περισσότερο τη σκέψη μου στη συνέχεια. Επίσης θα σας εξηγήσω πώς το ερωτηματολόγιο των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιείται ως πηγή πληροφοριών και ανάπτυξης δυνατοτήτων. Θα σας δώσω επίσης πληροφορίες σχετικά με το πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων. Ξεκινώντας λοιπόν από την ε, διαδικασία βασικές αρχές της διαδικασίας αυτής, η οποία είναι αρκετά πολύπλοκη, ξεκινάει από την ε, σταθεροποίηση των δυνατοτήτων, την, τον εντοπισμό δυνατοτήτων και με την ανάπτυξη των δυνατοτήτων. Η διαδικασία αυτή αποτελείται από δύο βασικές αρχές. Τον σχεδιασμό δυνατοτήτων και την υλοποίηση των δυνατοτήτων. Εμείς στο επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στρατιωτικό επιτελείο, είμαστε υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό δυνατοτήτων Η διαδικασία αυτή είναι ένας πρωταρχικός στόχος. Συγκρίνοντας τις α, στρατιωτικές προϋποθέσεις σε σχέση με το τι χρειαζόμαστε, τα κράτη-μέλη, σε ό,τι αφορά τις συμβολές τους, με άλλα λόγια συγκρίνοντας τι χρειαζόμαστε με το τι έχουμε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα. Κάτι το οποίο ανταποκρίνεται στην αναφορά πρόοδων. μετά τον εντοπισμό του ελλείμματος αυτού βλέπουμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι που προκύπτουν και αυτό είναι η λεγόμενη δύναμη A του σχεδίου. Το δεύτερο μέρος έχει να κάνει με την κατονόμαση των δυνατοτήτων και τη διευκόλυνση της ανάπτυξή τους. Το σχέδιο ανάπτυξης δυνατοτήτων κατευθύνεται από την Στρατιωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δυνατότητες αυτές είναι στρατιωτικά προϊόντα. Οι δυνάμεις A και D αποτελούν κομμάτι του σχεδίου ανάπτυξης δυνατοτήτων. Σε ό,τι αφορά τις συνεισφορές τώρα των κρατών μελών, Αυτές είναι σε εθελοντική βάση και οργανισμοί όπως ο Οργανισμός ε, Άμυνας της Υπηρεσίας Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να βασίζονται στις συνεισφορές αυτές. Πρακτικά τώρα, σε ό,τι αφορά τις δυνάμεις αυτές που χρησιμοποιούμε για την ανάπτυξη δυνατοτήτων, πρώτα απ' όλα είναι ανάγκη να εντοπίσουμε τη διαφορά ανάμεσα στο τι έχουμε και στο τι χρειαζόμαστε και η δύναμη D έχει να κάνει με τις δυνατότητες. Οι δυνάμεις C and B Το C αφορά στο τρέχον σχέδιο και το B έχει να κάνει με το μελλοντικό σχέδιο ανάπτυξη δυνατοτήτων για μελλοντικέ επιχειρήσεις μακροπρόθεσμα, οι οποίε αυτή τη στιγμή προβλέπονται για το 2025. Το ερωτηματολόγιο τώρα. Αποστέλλεται στα κράτη-μέλη. Μέχρι στιγμής είχαμε 17 απαντήσεις από τα κράτη-μέλη. Και θέλω να υπογραμμίσω ότι σε ό,τι αφορά το ερωτηματολόγιο αυτό έχει ένα χρονολόγιο το οποίο είναι απολύτως συγχρονισμένο με, την, με το σχεδιασμό και τη διαδικασία του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι και η αξία του. Δεν προσπαθούμε να κάνουμε ακριβώς αυτό που κάνει το ΝΑΤΟ. συμπληρωνόμαστε. Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε είναι διεξοδικές, αξιολογούνται και τίθενται σε σειρά προτεραιότητας. Όταν η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται, καταλήγουμε στο τμήμα A. Πώς ακριβώς λειτουργεί. Ε, επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα α, παράδειγμα ελλείψεων. Σε ό,τι αφορά τον ανεφοδιασμό αέρος, δεν μας επιτρέπει να επιχειρούμε να αέριες εκστρατείες. Τα αεροσκάφη λοιπόν που αποστέλλονται σε μακρινές περιοχές είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε την δυνατότητα ανεφοδιασμού στον αέρα προκειμένου να μπορούμε να επιτύχουμε τις επιχειρήσεις μας. Επομένως η αδυναμία του να έχουμε αυτή τη δυνατότητα είναι συνεπάγεται έναν τεράστιο επιχειρησιακό κίνδυνο. Ο ανεφοδιασμός αέρος είναι ένα σημαντικό ζήτημα ασφαλείας και είναι μια προτεραιότητα στο σχέδιο ανάπτυξης ικανοτήτων, δυνατοτήτων. Σε ό,τι αφορά τώρα το, το κομμάτι D, εδώ πρόκειται για ένα τομέα που αφορά στα μαθήματα που έχουμε μάθει. Και εδώ καλύγουμε καλύπτουμε πολλούς διαφορετικούς τομείς σε ό,τι αφορά τη σύνδεση, τα δόγματα, τη βιωσιμότητα. Πρώτα απ' όλα, στον τομέα αυτό μπορεί να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι χρειαζόμαστε κι άλλες δυνατότητες. Όταν αναπτύσσουμε τον τομέα Α, δεν διαπιστώσαμε ότι ο τομέας που αφορά στην καταπολέμηση των εκρηκτικών μηχανισμών έχει ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης κάτι το οποίο πιστοποιήθηκε και στους τομείς B and C. Σε ό,τι αφορά τα τρέχοντα θέματα, το που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά το σχέδιο ανάπτυξη δυνατοτήτων, αυτή τη στιγμή λαμβάνουν χώρα δύο παράλληλες διαδικασίες. Πρώτα απ' όλα, οι καινούριε στρατιωτικές προϋποθέσεις, έτσι όπως προκύπτουν από την Παγκόσμια Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάπτυξη των προϋποθέσεων αυτών προκύπτουν από ενδελεχή σενάρια που αφορούν σε δυνητικές επιχειρήσεις των στρατιωτικών επιχειρήσεων αλλά και ανθρωπιστικής βοήθειας. Βασιζόμενοι σε αυτό εντοπίζουμε τις διάφορες προϋποθέσεις, η διαδικασία είναι συνεχής. Όπως είπα, το ερωτηματολόγιο, το στρατιωτικό ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη αποσταλεί. Σιγά σιγά λαμβάνουμε απαντήσεις, πληροφορίες, feedback από τα κράτη-μέλη. Βεβαίως και όλες οι πληροφορίες για τις δυνατότητες επιχειρήσεων που λαμβάνουν χώρα. Τέλος, περνάμε στα συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα, οι νέες προϋποθέσεις, έτσι όπως προκύπτουν από την παγκόσμια στρατηγική, εξετάζονται και ένας καινούριο κατάλογος θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Δευτερευόντως, η τρέχουσα μεθοδολογία, τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να καταστήσουμε τον κατάλογο αυτό, είναι διαλειτουργικό με το ΝΑΤΟ. Στον τομέα λοιπόν αυτό, σε ό,τι αφορά το λογισμικό, για παράδειγμα, με άλλα λόγια, όταν εξετάζουμε πόσο πραγματικό είναι αυτό το οποίο προτείνουμε, μπορούμε να έχουμε καλύτερα συμπεράσματα. Σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις δυνατοτήτων, πρέπει να έχουμε την πλήρη, την πλήρη στήριξη των μελών, αλλά και τη βοηθειά τους για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων αυτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πριν δώσω το λόγο στους συντονιστές, και στα άλλα μέλη. Να θέσω και εγώ τα δικά μου ερωτήματα. Να αναφερθώ σε ασκήσεις ευρετικών απειλών. Είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν και οι εταίροι προς Ανατολάς, οι συνδεδεμένοι δηλαδή εταίροι, όπως για παράδειγμα πρώτη και καλύτερη Ουκρανία, μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει τις πιο υψηλές υβριδικές απειλές από πλευρά του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει και η συμφωνία πλαίσιο με το EDA και άλλες συμφωνίες που συμπληρώνουν τη συμφωνία ένταση και η CSTP. Η Ουκρανία, Μολδαβία μπορούν να συμπεριληφθούν λοιπόν αυτές οι δύο χώρες στις ασκήσεις αυτές. Πρώτο συντονίστης, ο κύριος Γκάλερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε και για τις δύο παρουσιάσεις. Χαίρομαι που βλέπω ότι η δουλειά σας συντονίζεται με όσα Πάντα δεν δεδεινόμαστε ότι χρειαζόμαστε και είμαι ευγνώμων για την ενημέρωση αυτή. Για όσο μας παρουσιάσατε. Μια συγκεκριμένη ερώτηση τώρα να σας κάνω για το σχέδιο δράσης. Έχουμε και το θέμα της έρευνας. Η συμφωνία αντιπροσωπείας μεταξύ της Κομισιόν και της ΕΝΤΑΣ υπογράφει τον Μάιο. Εξ όσων ακούω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Μαλλινομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει αναστείλει τις διαδικασίες. Για ενημερώστε με. Γιατί είχα την ελπίδα ότι θα είχε υπάρξει το πολιτικό πρόγραμμα και εκεί είχαμε επίσης ανάλογες ασκήσεις Ελπίζαμε λοιπόν ότι θα υπήρχε μια συμφωνία. Πού βρισκόμαστε. Στις 5.30 δυστυχώς θα πρέπει να προτρέψω μια άλλη συνάντηση, αλλά ο συνοδελφός μου θα μαζέψει τις απαντήσεις. Ο συνοδελφός Τρογεύσκη λοιπόν θα μαζέψει τις απαντήσεις σε περίπτωση που δεν προλάβω να, ακούσω την απάντησή Σα Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος, και να σα υπενθυμίσω ότι μεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μα και πάντα μπορούμε να ακούσουμε το περιεχόμενο της συνεδρίασή και των υστέρων. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λόζινγκ είναι η επόμενη Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή αυτή. Ω κοινή θνητή που δεν ε, κατανοεί απόλυτα τα θέματα των στρατιωτικών ικανοτήτων, πάντα με δυσκολεύει να δώσω μια συγκεκριμένη διάσταση σε όλα αυτά τα ζητήματα και να φανταστώ ποια συγκεκριμένα μέτρα προγραμματίζονται, κυρία Μορκερίνη. Προσπάθησα να το κάνω αυτό πιο συγκεκριμένο στους στόχους ε, τίτλους. Υπάρχει μια γενική διατύπωση κάποιων γενικών ε, ελλημάτων. Γι' αυτό λοιπόν ρωτώ κατά πόσον υπάρχουν συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία για ποιες ικανότητες συγκεκριμένα και ποιες δαπάνες εφαρμογής των ικανότητων αυτών χρειαζόμαστε. Άλλη μια συγκεκριμένη ερώτηση το CDP. Πότε θα προσαρμοστεί στο νέο σχέδιο ε, δράσεις, συμφωνώ με τον προλαλήσαντα. Και πώς εκτιμάτε την πιθανότητα να καλυφθούν τα κενά αυτά ικανοτήτων τα οποία μας παρουσιάσατε στην τρέχουσα παρουσίαση από το παράθυρο αυτό ικανοτήτων από το σχέδιο δράσης για την άμυνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Σκούζο. Δεν έχει σχόλια. Mr. Zdrojewski. Ε, κύριε Στροσχεύσκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια ερώτηση έχω να κάνω προς τον κύριο Λοιπόν, Ναύαρχο, μη σας πω και δύο ερωτήσεις. Πρώτον, γνωρίζουμε ότι το ΝΑΤΟ κάνει διαπραγματεύσει και θα έχει και μάλιστα παρατηρητέ ε, κατά πάσα πιθανότητα στις πιο σημαντικές, ε, στους πιο σημαντικούς ολιγμούς στη Λευκορωσία το Σεπτέμβριο του φετινού έτους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το στρατιωτικό επιτελείο θα προσπαθήσει να έχει καθεστώς παρατηρητή σε αυτά τα μεγάλα, σε αυτούς τους μεγάλους ολιγμούς, σε αυτές τις μεγάλες ασκήσεις στη Λευκορωσία. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση. Θα ληφθούν υπόψη και τα ζητήματα αυτά στην, στον υπολογισμό των ικανοτήτων. Σκοπεύετε να αξιοποιήσετε με διαφορετικό τρόπο το Ευρωπαϊκό αυτό σώμα προκειμένου να μπορέσει να εκτελέσει και άλλα καθήκοντα. Άλλη μια ερώτηση τώρα, επιτρέψτε μου προς τον, Α, στον υπονάβαρχο πάλι. Θα είσαστε διατεθειμένοι να πείσετε τον Πολωνό Υπουργό Άμυνας να μην ε, αποσυρθεί από το Ευρωπαϊκό αυτό σώμα. η Πολωνία θα έπρεπε να λάβει την ηγεσία του ευρωπαϊκού αυτού επιτελείου. Θα ήσασταν λοιπόν σε θέση και θα ήσασταν εντεθειμένος να δραστηριοποιείτε προς την κατεύθυνση αυτή. Μάλιστα, λέει η Πρόεδρος. Κύριε. Κύριε Διευθυντά, κύριε Υπονάμαρχε, παρακαλώ απαντήστε στα ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε οι υβριδικές ε, απειλές και οι σχετικέ ασκήσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας πω ότι κάνουμε δύο είδους ασκήσεις. Η πρώτη είναι πολυεπίπεδη άσκηση, η οποία έχει να κάνει με τη διαχείριση των κρίσεων σε υψηλό επίπεδο, με κάποια συμμετοχή του στρατιωτικού επιτελείου. Στην προκειμένη περίπτωση θα ήταν η κατάλληλη ευκαιρία να θέσουμε την υβριδική διάσταση πρακτικά όταν μιλάμε για τα υβριδικά ζητήματα. Κοιτάμε λιγότερο το σχετικό σκέλος και κυρίως τα άλλα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται για τέτοιου είδους υβριδικά σενάρια. Ως εκ τούτου, προφανώς εξαρτάται από τους υπεύθυνους δεν είμαστε εμεί αυτοί που διοργανώνουμε την άσκηση στην προκειμένη περίπτωση. Προσκαλούμε του συμμετέχοντε ως παρατηρητέ στις δικές μας ασκήσεις. Την Ουκρανία, τη Γεωργία, που παρατηρούν τις ασκήσεις αυτές. Με καθεστώ απλού παρατηρητή. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ξέρω ότι η παρουσίασή μου ήταν κάπως ακαδημαϊκή, αλλά νομίζω ότι δίνει μια ιδέα για το πώς έχει η διαδικασία. Και καλό θα ήταν ενδεχομένω σε ό,τι αφορά την παρουσίαση να ξεκινούσαμε με τον εντοπισμό των ε, προδιαγραφών, των αναγκών από πλευράς στρατιωτικής και μετά να κοιτάξουμε, να κοιτούσαμε πώς θα μπορούσαμε να να καλύψουμε τα κενά. Αυτό είναι πιο πολύ το σκέλος της ΕΝΤΑ. Πρακτικός πώς όμως. Να πω το εξή. Σε ό,τι αφορά τις, τα κρίσιμα, τις κρίσιμες ελλείψεις της ασκήσης, 14 έχουν εντοπιστεί από τις 42 στο σύνολο ελλείψεις. έχει να κάνει πιο πολύ με τα αριθμητικά στοιχεία. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις κρίσιμες αυτές ελλείψεις, τα κρίσιμα αυτά ζητήματα, προβλήματα, σε ό,τι αφορά την εποπτεία, τις μυστικές υπηρεσίες, τα στρατηγικά ζητήματα, τα διάφορα είδη αεροσκαφών. Μας λείπουν 650 για να καταλάβετε τα αριθμητικά στοιχεία. Όταν μιλάμε για ελλείψεις, ελλείμματα στις ικανότητές μας, για πραγματικά ελλείμματα αεροσκαφών για παράδειγμα. Να σας αναφέρω ότι ένα από τα προβλήματα και από τα ελλείμματα που έχουμε εντοπίσει είναι ο εντοπισμός, η ε, ταυτοποίηση και η ανείχνευση των δυνάμεων των αντιπάλων. Αυτό θεωρείται κρίσιμη, κρίσιμο έλλειμμα, κρίσιμη έλλειψη σε λειτουργικό επίπεδο. Τι σημαίνει αυτό σε επίπεδο συσκευών. Μιλάμε για 58 ε, αεροσκάφη αεροσδάφους. Μιλάμε για αεροσκάφη φυσικής υπογραφής, μιλάμε για ε, μονάδες ε, τηλεόρασης, IVU κτλ. Έτσι μεταφράζεται η έλλειψη ικανοτήτων σε πρακτικό επίπεδο συσκευών που μας λείπουν. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Τα λέω αυτά. Τώρα, για το... Να περάσουμε στην ερώτηση του Υπουργού Στοβιέσκη για το πρώτο ζήτημα το οποίο έθεσε. Για να σας πω την αλήθεια, δεν το σκεφτήκαμε. Δεν σκεφτήκαμε την άσκηση στην Λευκορωσία. Νομίζω δε ότι αναφέρθηκε το θέμα της της κοινή ε, κατανομής της ευθύνης και των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων και τη συμπληρωματικότητα σε ό,τι αφορά τέτοιε ασκήσει. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, είναι υπεύθυνη τόσο πολύ στην προάσπιση της ε, πατρίδος. Ε, είμαστε εστιασμένοι πιο πολύ στο εξωτερικό σκέλος και στην προκειμένη περίπτωση συμμετέχουμε στην διαχείριση της κρίσης για τις αποστολές εκτός τη Ευρωπαϊκής Ένωση και επίσης πιστεύω βλέποντας και την συμμετοχή στην Ουκρανία σε ό,τι αφορά το σταθετικό σκέλος δεν υπάρχει τέτοια συμμετοχή. Φυσικά θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε, θα μπορούσαμε να το θέσουμε σε πολιτικό επίπεδο αυτό το θέμα, το πώς δηλαδή και αν θα θέλαμε να συμμετέχουμε στην παρατήρηση, ως παρατηρητές μάλλον στην άσκηση της Λευκορωσίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό αυτό. Και το Eurocorp. Είναι ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, προφανώ. Το λέει και η λέξη. Αλλά δεν είναι το εργαλείο το οποίο είναι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχικά έχει σχεδιαστεί ως μία μονάδα η οποία θα υποστηρίζει βασικά τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πρακτική άποψη τώρα είναι διχασμένο. Και να σας πω, το Στρατιωτικό Επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει υπογράψει επιστολή προθέσεων και υπάρχει και μια σχετική ομάδα εργασία η οποία ιδρύθηκε και έχει εντοπίσει τομεί στους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Επιτελείο και το Eurocorp θα μπορούσαν να συνεργαστούν. Το Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Επιτελείο είναι σε επαφή με το Ευρωπαϊκό αυτό σώμα, το Eurocore, σε τακτική βάση. Και βραχυπρόθεσμα θεωρώ ότι θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Eurocore. Γιατί υπάρχουν επιπρόσθετε πλέον δραστηριότητε στο στρατιωτικό επιτελείο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναπτύσσουμε το διοργανωτικό σκέλο user planning conduct capability. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει αφιερώνεται για την ε, εφαρμογή αποστολών μη εκτελεστικής φύσης. Για παράδειγμα στην Αφρική, το Eurocore ε, έχει ηγετική θέση ο επικεφαλής, είναι από το Eurocore και ένα μεγάλο τμήμα του επιτελείου είναι από το Eurocore. Έτσι έχει η κατάσταση σήμερα, εκ παραλίλου. Βάσει και των συναντήσεων που έχουμε κάνει με την ηγεσία του Eurocore, λαμβάνουμε τις πληροφορίες ότι τα επόμενα δύο έτη το Eurocore θα επικεντρωθεί στο ΝΑΤΟ. Αυτό τι σημαίνει ότι η συνεργασία του Eurocore με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι περιορισμένη. Έτσι έχουν τα πράγματα με το Eurocore. Πρακτικά τώρα σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της Πολωνίας στο Eurocore. Νομίζω ότι κατανοείτε ότι το θέμα αυτό είναι αμυγός πολιτικό. Γι' αυτό λυπάμαι, αλλά δεν θα το σχολιάσω. Δεν θα σχολιάσω το ποια θα είναι η πλέον ενδεδειγμένη κατεύθυνση να ακολουθηθεί. Αυτά είχα να σχολιάσω. Ευχαριστώ. Bardzo dziękuję Pani Admirale. Now I like to... Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Γκος. Καταρχήν να απαντήσω στη δική σας ερώτηση σε ό,τι αφορά την άσκηση επιχάρτου για τις υπηρετικές απειλές. Έχουμε μια, κάποιες διοικητικές διευθετήσεις όχι μόνο, για την, όχι μόνο με την Ουκρανία αλλά και με την Ορβηγία, την Ελβετία, τη Σερβία και την Ουκρανία. Σε ό,τι αφορά τις ασκήσεις η Ουκρανία δεν είχε προσκληθεί αλλά αν θυμάμαι καλά Δεν, είχαμε, δεν θυμάμαι καν αν είχαμε διοικητικέ διευθετήσει με την Ουκρανία. Δεύτερον, για να προσκληθούν χώρες μη μέλη στις δυτικές αυτές διευθετήσεις χρειάζεται ομοφωνία των μελών. Προφανώ δεν είναι πρόβλημα, αλλά αυτή είναι η διαδικασία. Και αυτή η διαδικασία θα εφαρμοστεί και στο μέλλον, προκειμένου να προσκληθεί η Ουκρανία, αν είναι δυνατόν. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ερώτηση Γκάλος. Χαίρομαι που θεωρείτε πως η δουλειά είναι, απαντά στις ανάγκες σας. Σε ό,τι αφορά την ΕΔΕΠ, ε, θα έπρεπε να έχει υπογραφεί αρχές Μαΐου. Τώρα στόχος είναι ο Μάιος και πάλι, ίσως το τέλος Μαΐου. Είναι αλήθεια ότι το πιλωτικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε έγκαιρα, όχι όμως και χωρίς ε, ε, έντονες διαπραγματεύσεις και δύσκολες διαπραγματεύσεις. Εδώ έχουμε ακόμα περισσότερες, περισσότερους παράγοντες που εμπλέκονται, νομικούς και άλλους. Ελπίζω και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα είμαστε έτοιμοι έγκαιρα. Ήδη προετοιμαζόμαστε Έχουμε στελεχώσει την, ε, ε, το τμήμα ε, δράσεων προετοιμασίας και νομίζω ότι όλα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Τρίτον, κύριε Λέζινγκ, θα, θα μιλήσω λίγο γερμανικά αν μου επιτρέπετε. Είπε προτιμάτε αγγλικά. Ε, μιλήσατε για κενά στρατιωτικών δυνατοτήτων και τι μέτρα παίρνουμε για να τα πληρώσουμε. έχω μια εύκολη απάντηση, απλή απάντηση, που δεν είναι όμως σωστή απάντηση. Ε, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εμείς μέσω του CDP ε, δίνουμε στα κράτη-μέλη μαζί με την βάση δεδομένων συνεργασίας που διαθέτουμε, κονταμπά, έτσι λέγεται, κονταμπά, ε, δίνουμε στα κράτη-μέλη την εικόνα για το πού βρισκόμαστε, τι ευκαιρίες έχουν, τι ανάγκες υπάρχουν κλπ. Ε, εκεί που υφίστανται αδυναμίες το θα το δουν τα κρατη και θα κάνουν τον προγραμματισμό τους, τριετή, πενταετή κλπ. Για παράδειγμα, μία πανδρομένα αεροσκάφη, ε, ε, πλοία, σκάφη κλπ. Θα δούμε λοιπόν ότι για παράδειγμα 9-10 κράτη-μέλη μπορεί να έχουν τις ίδιες ανάγκες και θα τους πούμε γιατί δεν έρχεστε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας να εναρμονίσουμε αυτές τις ανάγκες και έτσι θα διευκολύνουμε ένα πρόγραμμα αγοράς ε, προμηθειών για παράδειγμα αεροσκαφών που ανεφοδιάζονται στον αέρα. Ε, και έχουμε τα κράτη-μέλη λοιπόν που ε, είναι η κινητήρια δύναμη ε, και υπάρχει μια παροιμία που λέμε μπορούμε να πάμε το άλογο να πιει νερό αλλά δεν μπορούμε να το αναγκάσουμε να το πιει. Έτσι κάνουμε και εμείς. Εμείς διευκολύνουμε τα κράτη-μέλη αλλά τα κράτη-μέλη τελικά θα αποφασίσουν. Σε ό,τι αφορά το κόστος. Και αυτό εξαρτάται από το εθνικό, από τα εθνικά σχέδια προμηθειών. Εμείς ε, ζωγραφίζουμε την εικόνα, ε, εντοπίζουμε τις αδυναμίες, τα κενά κλπ. Αλλά τελικά δεν θα αποφασίσουμε εμείς τι θα κάνει το κάθε κράτος μέλος. Δίνουμε τον πίνακα στα κράτη-μέλη και ελπίζουμε ότι θα τον διαβάσουν καλά, θα τον παρατηρήσουν και θα ε, ενταχθούν σε κοινά προγράμματα. Τριών, τεσσάρων, πέντε κρατών ή και πιο πλατιά και ευρεία συμμετοχή όπω ο ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό που συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη. Αυτέ νομίζω ήταν οι ερωτήσει που αφηθήθηκαν σε μένα. Ε, Κύριε Στογεύσκη, Ε, αλλαγή στο Eurocore σημαίνει ενδεχομένω και αλλαγή στον εξοπλισμό του πιστεύω ότι στο CDP θα, από το CDP θα γίνει εμφανές ότι ε, το κάθε κράτος μέλος θα έχει τις δικές του ανάγκες. Πριν από πέντε χρόνια, για παράδειγμα, πολλά κράτη-μελή είχαν πει, σκεφτόντουσαν ότι δεν χρειάζονται πια τάγκ. Βλέπετε όμως ποιο είναι το αποτέλεσμα σήμερα. Πολλά κράτη-μέλη χρειάζονται περισσότερα τάγκ. Και αυτό μπορεί να ισχύει και σε άλλου τομεί, όπω για παράδειγμα συλλογή πληροφοριών, παρακολούθηση και επιτήρηση. Και με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε και την συνεργασία των κρατών μάλλον καλύτερα, να κάνουμε περισσότερα και περισσότερα πράγματα μαζί. Indeed, uh, there is still time Υπάρχει χρόνος για περαιτέρω συζήτηση. Βλέπω όμως ότι δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας ημερήσια διάταξη και θα ήθελα να ευχαριστήσω τα αξιότιμα μέλη του πάνελ μας για τις παρουσιάσεις τους. σε ό,τι αφορά το CDP και την αναθεώρησή του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη για τη συμμετοχή τους στη συζήτηση. Έπειτα από ένα εξοντοτικό πρώτο μέρος της σημερινή συνάντησης και επίσης να σας υπενθυμίσω ότι αύριο υπάρχει μια αλλαγή σε ό,τι αφορά την αίθουσα που θα συναντηθούμε. Θα ξεκινήσουμε στις 9 και το νούμερο της αίθουσας είναι π485. 011. Οπότε παρακαλώ σημειώστε την αλλαγή αυτή στην αίθουσα. Σας ευχαριστώ και πάλι κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ κύριε Διευθύντα. Σας παρακαλώ πολύ ένα θερμό χειροκρότημα για τους ομιλητές μας.